Κυρίες και κύριοι, το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι η προφορική ερώτηση προς την ε, Επιτροπή για την Ελεύθερη Κυκλοφορία Εργαζομένων προσωρινή περιορισμή που αφορούν Ρουμάνους και Βούλγαρους πολίτες στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς να δώσουμε το λόγο για να διατυπώσει την ερώτηση στην κυρία Πλάμπ. Uh, Κύριε Πρόεδρε,